Η διάταξη βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς για την ευελιξία τους και διάθεσή τους. Πέρα στη συζήτηση.